Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτηση που αφορά τη Συρία. Αλλά πριν ε, είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπατε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Εξωτερικέ Υποθέσει και την Πολιτική Ασφαλεία, την κυρία Μογκερίνη, η οποία εν συντομία θα μα μιλήσει για δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσει για την πρόοδο όσον αφορά το σύμφωνο του ΟΗΕ που αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ούτω ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε νόμιμη μετανάστευση υπό συνθήκες ασφαλεία και τάξεως και δεύτερον οι προπτικές για ειρήνη για την κορεατική ε, Χερσόνησο υπό το φω των προσφάτων ε, γεγονότων και εξελίξεων. Έτσι λοιπόν η κυρία Αντιπρόεδρε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το Παγκόσμιο Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την με, για, τους μετανάστες, για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες να ξεκινήσω με μία επιτέλους χαρμόσυνη είδηση. Και είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ευρωπαϊκό επίτευγμα των τελευταίων μηνών. Θα θυμάστε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο είχα έρθει στο Στρασβούργο, εδώ στην Ολομέλεια, και μιλήσαμε για τα κέντρα κράτησης ε, στη Λιβύη. Και μάλιστα είχα αναλάβει ενώπιον σας και ενώπιον ε, όλων ε, όσων υφίσταται τα πάνδυνα στα κέντρα κράτης της Λιβύης να ε, επιστρέψουν 15.000 μετανάστες από τα κέντρα αυτά στις α, ε, χώρες προέλευσής τους με ασφαλή τρόπο και με το σύστημα εκούσιας επιστροφής που διαχειριστήκαμε από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετανάστευση. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία άνευ προηγουμένου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Αφρικανική Ένωση και ε, με τι υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών για μετανάστες και πρόσφυγε στην διάσκεψη κορυφής του Αμπιτζάν που έγινε με την Αφρικανική Ένωση. Και χάρη στη συμφωνία αυτή, τους δύο πρώτους μήνες του 2018, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, καταφέραμε να διασώσουμε και να απελευθερώσουμε πάνω από 16.000 ανθρώπους από, τα, από τους καταβλισμούς προσφύγων στη Λιβύη. Και μέσα σε δύο μήνες καταφέραμε όσα είχαμε καταφέρει τον προηγούμενο, ολόκληρο τον προηγούμενο χώρο. Και το 2017 ήταν δεκαπλάσια, δέκα φορές καλύτερα τα αποτελέσματα από ό,τι το 2016. Και τώρα στα κέντρα κράτησης, στους καταβλισμούς προσφύγων έχουν απομείνει 4 με 5.000 ε, άνθρωποι. Παρά είναι μεγάλος αριθμός και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, αποκοινούμε τα Ηνωμένα Έθνη της, ε, και την Αφρικανική Ένωση να εκενωθούν ε, αυτά τα στρατόπεδα, αυτά, αυτοί οι καταβλισμοί και μια και σε δύο μήνες καταφέραμε να απελευθερώσουμε 16.000 φαντάζομαι τους επόμενους μήνες θα καταφέρουμε να απελευθερώσουμε και τους υπόλοιπους. Και αυτό κατέστη δυνατό κυρίως για ένα λόγο. Συσπυρώσαμε τις δυνάμεις μας, κυρίως εντός της Ευρώπης και σε συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους και φίλους αλλά και παγκοσμίω στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Και ξεκινώ με αυτή τη θετική νότα, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι πολύ δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε να εστιαστούμε στα επιτεύγματα, στα θετικά σημεία και είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και τα θετικά, τα επιτεύγματά μας, γιατί αυτά θα μας καθοδηγήσουν στις υπόλοιπε λύσεις. Βέβαια αυτό είναι μόνο μια ψηφίδα του ψηφιδωτού που προσπαθούμε να συστήσουμε. Θέλουμε ε, ένα, μια μέθοδο ασφαλών και εξωπρεπών επιστροπών και διάσωση ζώων και χερσαία και στη θάλασσα. Επίσης να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της μετανάστευσης και με το νέο εξωτερικό ταμείο να δημιουργήσουμε ε, ανάπτυξη και απασχόληση και στις χώρες της Αφρικής. Τεράστιες οι προκλήσεις βέβαια και έχουμε τις έχουμε βιώσει και εμείς, αλλά οι Αφρικανικοί και άλλες ήπειροι βιώνουν τις προκλήσεις αυτές ακόμη πιο έντονα. Βέβαια, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, όχι από καμία χώρα μόνη της, αλλά με συνεργασία για να έχουμε έναν πραγματικά αξιοπρεπή μηχανισμό για να διαχειριστούμε την παγκόσμια κινητικότητα. Και μάλιστα πριν από δύο χρόνια αποφασίσαμε για την αλληλεγγύη, την κοινή ευθύνη, την πολυμέρεια και τη δέσμευση. Αυτοί είναι οι τέσσερις πυλώνες που συνιστούν το κοινό έδαφος της συνεργασίας μας και επίσης ε, διέπουν και τα δύο παγκόσμια σύμφωνα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Δεν είναι μένοντα απλέ παρατηρητές, ή χτίζοντα τύχη μεταξύ μόνο και του υπόλοιπου κόσμου που θα, θα, θα βρούμε κοινέ λύσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλες οι χώρες θα υποφεληθούν από στενή ε, παγκόσμια συνεργασία και οι χώρες προέλευσης και διέλευσης και προορισμού. Και μάλιστα μερικές χώρες ε, έχουν και τα τρία χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι και χώρες προέλευσης αλλά και ταυτόχρονα χώρες διέλευσης και προορισμού. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις εργασίες και στα δύο παγκόσμια σύμφωνα ε, οι διαπραγματεύσει και οι επίσημε διαβουλεύσει ξεκίνησαν για το κείμενο τον περασμένο μήνα και νομίζω ότι έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό όραμα για τη μετανάστευση. Και μάλιστα να το αναγάγουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και να μεταφέρουμε τι εμπειρίε μα, τα διδάγματά μα και τι εταιρικέ σχέσει που δημιουργήσουμε. Ένα όραμα που θα δράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ευθύνη και στην αμοιβαία αλληλεγγύη. Ένα όραμα που οι λαθροδιακινητέ, οι λαθρέμποροι και τα εγκληματικά κυκλώματα δεν θα έχουν θέση. Θα μειώσουμε την παράτυπη μετανάστευση και ταυτόχρονα θα έχουμε το θάρρος να επενδύσουμε σε πιο νόμιμες οδούς για τους μετανάστες. Και θέλουμε στενή συνεργασία στα Ηνωμένα Έθνη ε, υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετανάστευσης. Και μάλιστα ε, έχουμε πίσω μας τις πρώτες ε, διασκέψεις στη Νέα Υόρκη με μεγάλη συμφωνία αλλά πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας. Πάντως υπάρχει καλή βάση για να καταλήξουμε στη συνεννόηση, ώστε με ε, αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο να διαχειριστούμε και τώρα και μακροπρόθεσμα τη μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο για του Πρόσφυγε, ήδη έχουν ξεκινήσει επίσημε διαπραγματεύσει στη Γενέβη. Θέλουμε μια ισορροπημένη ε, έκβαση και για του πρόσφυγε και για τις ε, κοινότητε που του υποδέχονται τους τελευταίους 18 μήνες ε, πρωτοστατήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαδικασία αυτή, χάρη και σε εταιρικέ σχέσεις που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια. Και τώρα με την αποχώρηση από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια ε, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη. Και μάλιστα δυστυχώ ε, ένα κράτο μέλο πρόσφατα παρουσίασε μια θέση που δεν ευθυγραμμίζεται με τη θέση των υπόλοιπων 27 χωρών. Και εδώ το κοινό μα έργο, αλλά και η δική σα συμβολή, η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει μεγάλη σημασία. Γιατί από κοινού μπορούμε να προωθήσουμε ε, ισορροπημένα σύμφωνα, χωρί αποκλεισμού, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, να καλύψουμε τι συμφωνίε των Ευρωπαίων πολιτών και να μετατρέψουμε την μετανάστευση από, από πρόκληση σε κοινή ευκαιρία. Τώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Περνάμε από τα Ηνωμένα Έθνη στην Κορεατική Χερσόνησο. Για μήνες και χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποφύγει το σενάριο του εφιάλτη μιας πυρηνικής κρίσης στην Κορεατική Χερσόνησο. Γνωρίζετε ότι έχουμε αποκομίσει κάποια εμπειρία από το έργο μας σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Και μετά τους χειμερινού, με τους, Ολυμπιακούς, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς στην Κορέα και τώρα με τους Παραολυμπιακούς έχει διαμορφωθεί κάποιο διαφορετικό κλίμα. Και η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο μπορεί να μετατραπεί από μια δυνητική καταστροφή σε μία απόδειξη της ισχύω της πολυμερούς διπλωματίας και μιας σοφής ηγεσία. Και θα ήθελα εδώ να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω τις προσπάθειες της Κορεατικής Δημοκρατίας και του Πρόεδρου Μουν για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες η Βόρεια Κορέα ε, στόματος του ειδικού επεσταλμένου ε, έδειξε προθυμία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ε, για αποπυρηνικοποίηση. Και αν οι αγγελίε αυτέ ε, τη Βόρεια Κορέα υπεβεβαιωθούν, θα δημιουργήσουν τι απαραίτητε προποθέσει και πρόσφορο έδαφο για μία λύση που θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Το καλοκαίρι, μάλιστα την πρώτη συνάντηση του, ε, των ηγετών τη Βορείου και Νοτιού Κορέα ε, τον Απρίλιο, θα είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση τη σχέση. Και η πιθανή ετοιμότητα του Πρόεδρου Τραμπ να αποδεχθεί την πρόσκληση τη Σύνοδο Κορυφή του Μαΐου, ίσω αποτελέσει ένα επιπλέον στοιχείο μια ρηξικέλευθη ε, θετικής λύσης. Και φυσικά η θέση της παγκόσμιας κοινότητας θα είναι κέρια για να δούμε αν θα επιτύχουμε ή θα αποτύχουμε στη διαδικασία αυτή. Εμείς οι Ευρωπαίοι και τα κρατημέλη είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το δικό μας καθήκον όπως πάντα και να, να δεσμευτούμε και στη Βόρεια Κορέα ε, με κριτική βέβαια στάση ασκώντας και πίεση αλλά και ε, όντας θετική προς το διάλογο. Το βασικό είναι να αποτρέψουμε τον κίνδυνο του πολέμου και να καταλήξουμε σε μία αποπυρηνικοποίηση της κορατική χερσονήσου ε, μάλιστα χωρίς ε, δυνατότητα επαναφοράς σε πυρηνικοποίηση. Πάντως το καθεστώς τη Βορείου Κορέας είναι το πιο περιοριστικό στον κόσμο Εμεί έχουμε εφαρμόσει όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βόρεια Κορέα και έχουμε και αυτόνομα επιπλέον μέτρα. Και βοηθούμε και τρίτε χώρε να εφαρμόσουν πλήρω τα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και απευθύνουμε έκκληση προ τι τρίτε χώρε, διατηρώντας την άμεση και έμεση πίεση προ τη Βόρεια Κορέα. Πάντως θεωρούμε ότι οι κυρώσει δεν είναι αυτός σκοπό, αλλά μέσο, εργαλείο, στόχο ήταν είναι και θα είναι η διάνοιξη πολιτικής οδού για την ε, ανέβρεση λύσης ε, συνενετικής με τη Βόρεια Κορέα. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε τις νέες διπλωματικές ε, προσπάθειες υψηλού επίπεδου και θα ήθελα να χαιρετήσω την ηγεσία και το θάρρος του Πρόεδρου μου και της κυβέρνησης της Νοτιού Κορέας. Είμαι περιχαρής και υπερήφανα. Σας αναγγείλω την επόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες θα υποδεχθώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιοκορέας στο Συμβούλιο Εξωτερικών για να συζητήσουμε το μέλλον και το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Νότιου Κορέας ε, και τις προσπάθειές της, όπως κάναμε και τους τελευταίους μήνες και ελπίζοντας να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Στόχος μας, όπως είπα, είναι η πλήρης, ε, ελέγξιμη ε, και οριστική αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου. Και πιστεύω ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος αν επιδείξουμε σύνεση, σοφία, ενότητα και αποφασιστικότητα πυγμή, όπως κάναμε μέχρι στιγμής ε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.